διαδρομικών αναμεταδόσεων. Και θέλω να δώσω το λόγο αμέσω στον συντάξοντα, τον κύριο Φίσερ, για 5 λεπτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Η Επίτροπο Κρού δυστυχώ σήμερα δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Θα ήθελα να τη ευχηθώ περαστικά, γιατί ξέρω ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας. Πολιτικά δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί τη, ε, βλέποντας τι σχεδιάζει όσον αφορά τον τομέα αυτών των κρατικών ε, ε, υπηρεσιών, των δημοσίων υπηρεσιών, των διευθυντικών μεταδοσίων. Με την κυρία και άλλη μια οργάνωσα μια κρόση για το θέμα της ανακοίνωσης της Κομισιόν για το θέμα αυτό και μπορώ να σας ε, ε, πω ότι πραγματικά τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ακόμα και η Γενική Διεύθυνση Αναγωνισμού ε, είχε αποστείλει πολλούς συνεργάτες το θέμα είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό Ο Γενικός Διευθυντής του τομέα της, Αγωνισμού ήταν παρόν όλο το πρωί ε, πρόκειται δηλαδή εδώ για την προετοιμασία διατάξεων για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες ε, ραδιοτηλεοπτικής ε, αναμετάδοσης. Αυτό που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι αποδεκτό. Έχω πολλά να επικρίνω στα σχέδια αυτά. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ε, οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες είναι εθνικό θέμα. Τα εθνικά κράτη δηλαδή θα πρέπει να εργαστούν σωστά, όχι η Κομισιόν. Θα ήθελα να σας πω ότι τα κράτη-μέλη οργανώνουν και χρηματοδοτούν με το δικό τους τρόπο τους ε, δημόσιους υπηρεσίες ε, ε, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Εδώ η Κομισιόν δηλαδή διαταράσει την αρχή της επικουρικότητας. Πρόκειται για εθνικά μέτρα, για κοινοτικά μέτρα αντί για εθνικά μέτρα και αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου σωστό. Έχω λοιπόν πάρα πολύ σοβαρέ επιφυλάξει για την πρόταση αυτή, γιατί πρόκειται για μια αξιολόγηση εξάντε. Ε, Εδώ τι γίνεται, δημιουργείται συμπληρωματική γραφειοκρατία. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μικρές ε, οι υπηρεσίες έχουν την ε, επαρκή μέσα για να το κάνουν. Και ποιο θα πληρώσει. Ναι. Για μικρές χώρες κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτα. Αυτά τα τέσσερα είναι πολύ λεπτομερή, δεν υπάρχει καμία ευελιξία στην πρόταση. Το μόνο που θα γίνει θα είναι ότι τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτό που επιβάλλεται. Και τώρα η αξιολόγηση εξάντε των επιπτώσεων στην αγορά θα έχει κάποια αξία. Μήπως τελικά οι εμπορικοί σταθμοί θα είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν. Τρίτον, με ανησυχεί αυτή η πρόταση γιατί δεν είναι κατά τον τρόπο οργανωμένοι οι κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί, διαφορετικές οργανώσεις, χώρες διαφορετικού, ε, συγγνώμη, ε, εκπομπές διαφορετικού μεγέθους. Αυτά που προτείνονται αυτή τη στιγμή είναι στάνταρτ, είναι ε, λύσεις που πρόκειται να ταιριάσουν σε όλους. Αυτό δεν θα λειτουργήσει όμως. Αυτές είναι οι ησυχίες μου και να σας πω τώρα και ε, κάτι σχετικά με την ακρόαση της περασμένης Πέμπτης. Τώρα μας ακούτε. Υπάρχει πάρα πολύ... Είναι πολύ σημαντική δουλειά. Η Κομισιόν μου είπε ότι η οριστική ανακοινώση ίσως αναβληθεί μέχρι μετά τις 5 Μαρτίου, ε, Μαρτίου γιατί τότε η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων θα οργανώσει μια νέα ακρόαση και μετά την ακρόαση αυτή, είπε ο Γενικό Διευθυντή, η Κομισιόν βάσει των νέων πληροφοριών ίσω υποβάλει μια νέα, νέα πρόταση πριν υποβάλει την οριστική ανακοίνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα αυτό. Και γι' αυτό εξεπλάγει μια από αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν άνοιξε επιτέλους τα μάτια της και προτίθεται να ακούσει και το τομέα και το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό δεκτό. Έχω ορισμένε ερωτήσει προ την Κομισιόν. Πρώτον, η Κομισιόν ε, θα επιμείνει σε αυτό το λεπτομερή έλεγχο της αγοράς από ανεξάρτητες θέσεις. Σε αυτό θα μπορείτε να προωθήσετε προς την Επίτροπο ε, Κρούς. Θα επιμείνει η Κομισιόν ή δεν θα το κάνει, δεν θα έχει μια ανεξάρτητη επιτήρηση και έλεγχο της αγοράς. Κατόπιν, τεχνική ουδετερότητα. Πώς θα το εξασφαλίσετε αυτό. Το κείμενο που έχουμε εδώ ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σχετικά με τις παλιές και τις νέες ε, ε μορφές. Θα πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν επίση αν προτίθεται να υποβάλει νέα πρόταση μετά από νέε πληροφορίε. Τέταρτον, τι θα κάνει η Κομισιόν σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για την ε, δανεική υπηρεσία ΤΕΦΑ 2 και εάν όχι τι θα κάνει και πέμπτον προτίθεται η Κομισιόν να ε, δώσει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο Κοινοβούλιο στην προετοιμασία της πρότασής της. Εγώ ελπίζω να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και Κομισιόν και κρατών μελών για να έχουμε μια καλή ανακοίνωση του τέλους. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Πίτροπος. Uh, κυρία Πρόεδρε, όπως ήδη έχει λεχθεί η συνάδελφος κυρία Κρούζ είχε ένα μικρό ατύχημα γι' αυτό δεν είναι παρούσα εδώ. Στις 4 Νοεμβρίου 2008 η Κομισιόν δημοσιεύσε για διαβούλευση μέχρι την 8 Ιανουαρίου ένα κείμενο η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου έχει οργανώσει μια συζήτηση για τις 5 Μαρτίου και το ΕΛΚ ήδη έκανε μια ακρόαση την περασμένη πέμπτη ε, την παρουσία του κυρίου Φιλιπλό ο διάλογος κομισιών και για κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικός περιμένουμε να σας ακούσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2008 αποφάσισε ότι θα πρέπει να δίνεται μια κάποια κρατική βοήθεια σε κάποιους ε, οργανισμούς για να ε, επικοινωνιακούς τους ώστε να αποφεύγονται προβλήματα πολιτικής φύσεως και άλλα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δημόσια ε, ραδιοφωνία και τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ σημαντική ιδιαίτερα να δούμε την ε, πλατφόρμα των ΜΜΕ ε, και πραγματικά προσπαθούμε να και βελτιώσουμε την κατάσταση, να διατηρήσουμε τουλάχιστον την κατάσταση των κρατικών ε, επιδοτήσεων που ξεκίνησε με την ανακοίνωση το 2001. Εξυγχρονισμός της επικοινωνίας είναι ένας στόχος μας, αλλά με διαφάνεια και νομική ασφάλεια. Η... Το σχέδιο ανακοίνωσης λέει ότι οι δημόσιοι σταθμοί μπορούν να παράγουν, θα πρέπει μάλλον να παράγουν, να έχουν εκπομπές σε όλο το οπτικοακουστικό φάσμα και πλατφόρμα. Έτσι κι αλλιώς αυτό ε, διασφαλίζεται και με το κείμενο του Αμστερντάμ που ε, ρυθμίζεται σχετικά σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, το τεστ που γίνεται σε εθνικό επίπεδο ε, βοηθάει γιατί δεν επεμβαίνει η Κομισιόν παντού και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να υπάρχουν ορισμένα πράγματα για τα οποία να ενδιαφέρεται η αγορά αλλά το κοινό δεν ενδιαφέρεται. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ιδιαίτερα με αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις να παίρνονται αποφάσεις και να δίνονται λύσεις και εμείς σεβόμαστε εδώ την επικουρικότητα και δεν επεμβαίνουμε αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε τα πράγματα. Το τεστ του Αμστερνταμ πιστεύουμε ότι ικανοποιεί και τους θεατές και τους ακροατές ε, και ελαχιστοποιεί τις πιθανές βλάβες αν θέλετε που θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχουν για τους ιδιωτικούς φορείς δεν ε, συμφωνούμε ότι είναι πολύ δύσκολο το τεστ και υπερβολικό βεβαίως χρειάζονται προσπάθειες αλλά πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή το τεστ που γίνεται και το και από εκεί και πέρα υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πότε κάποιες νέες υπηρεσίες που παρέχονται χρειάζεται να ελεγχθούν, να δοκιμαστούν. Από οι δημόσιοι φορείς μπορούν από εκεί και πέρα να ε, πειραματίζονται με νέα μέσα χωρίς ε, προηγούμενο τεστ Επα, επίσης δίνεται πλήρης ελευθερία ε, και στους θεσμούς και ανεξαρτησία στους θεσμούς που εφαρμόζουν το τεστ τώρα από εκεί και πέρα το Βέλγιο και η Ιρλανδία όπως θα ξέρετε ήδη εφαρμόζουν το τεστ αυτό και οι λύσεις που βρέθηκαν στις χώρες αυτές είναι ανάλογες με τις ε, ε, οικονομικές δυνατότητες ε, το τεστ που δεν είναι λόγο περιορίζει την εδαφική ελευθερία ε, εκείνο που εξασφαλίζει είναι ότι καλύπτονται οι κοινωνικές και άλλες ανάγκες της κοινωνίας και επίσης για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των ε, ε, φορέων ε, Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δίνουν, τη διακριτική, δίνουν διακριτική ευχαίρεια για το τι θα γίνει στους ίδιους τους φορείς εκπομπών. Πιστεύουμε ότι το τεστ αυτό θα διατηρήσει τον πλουραλισμό στον χώρο των ΜΜΕ και, για τα, και θα βοηθήσει και τα εμπορικά μέσα και τις εφημερίδες online και τα Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στην, τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτον, από το ΕΛΚ, ο κύριος Μπέλετ. Έχει το λόγο για τρία λεπτά. Κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Κυρία Επίτροπε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση στην κυρία Κρούς. Προσβλέπουμε να την δούμε εδώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε καλή υγεία πάντα. Να προχωρήσω. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή θέλει να υπάρχει ισότιμη βάση λειτουργίας όλων των ε, υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτική ε, μετάδοσης, ιδιωτικών και δημησίων. Αυτό είναι κρίσιμο και χρειάζεται να υπάρχει και σωστό επίπεδο ποιότητας. Αυτό που θέσπισε, ε, που προτάθηκε από την Επιτροπή και αυτό που είπε η κυρία Φίσερ δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές αυτές πάντα. Το τεστ αγορά, όπως το προτείνεται εφαρμόστηκε εφαρμόστηκε ήδη στο Βέλγιο, είπατε. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Χρησιμοποιούμε ένα, μια αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, οι ίδιες οι εταιρείε, οι τα κανάλια το κάνουν, αλλά η εικόνα που αποκαλύπτεται δεν είναι αυτή ακριβώς που περιγράψετε. Να σας πω ποιες είναι οι ανησυχίες που έχουμε και εμείς και η ομάδα μας. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι έρχεται ε, κόντρα ακριβώ στην στρατηγική της Λισαβόνας. Οι δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόραση στα κράτη-μέλη ε, αποτελούν το κέντρο της ραδιοτηλεοπτική πολιτικής αλλά δεν έχουν το κέντρο των εσόδων. Στην πραγματικότητα ε, οι οργανισμοί αυτοί έχουν σοβαρή, σοβαρά προβλήματα γραφειοκρατικού και χαρακτήρα που δημιουργούν επιπλέον δαπάνες και οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να διασπαρούν όσο περισσότερο γίνεται εξασφαλίζοντας ότι και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς μαζί θα δημιουργήσουν τις νέες αυτές πλατφόρμες και κατόπιν θα προσφέρουν το περιεχόμενο των πλατφόρμων αυτών. Έτσι θα προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα στον καταναλωτή. Μην παρανοείτε ωστόσο, μην, μην παρανοήσετε αυτά που θέλουμε να πούμε. Εμεί θέλουμε να υπάρχει ισορροπημένος ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και πρέπει να υπάρχει χώρο και για τους δύο, ούτως ώστε και οι δύο να παράσχουν περιεχόμενο ποιοτικό. Και προφανώς οι δημόσιες επιχειρήσεις ραδιοτηλεόρασης θα πρέπει να στηρίζονται σε δημόσια κονδύλια. Αυτό είναι προφανές. Δεν νομίζω ωστόσο ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Αν μου επιτρέπετε να παραπέμψω και λίγο στο BBC. Αν δείτε την τις εξαιρετικές μεθόδους παραγωγής και διανομής που έχει καταφέρει να πετύχει το BBC, θα δείτε ότι αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπατζελή, τρία λεπτά για το, τη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασιλείου, σας εύχομαι καλή χρονιά, καθώς και στην κυρία Κρόες γρήγορη ανάρρωση κύριε επίτροπε αναθεώρηση των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στα δημόσια οπτικοακουστικά μέσα η οποία προωθήθηκε από τη γαλλική προεδρία αποτελεί μια εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση για το εσωτερικό πολλών κρατών όσο και για τη θέση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ταυτόχρονα όμως με την αναθεώρηση του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες όπου ουσιαστικά αναδιαρθρώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο τρόπος και τα κριτήρια διανομής του ραδιοφάσματος καταδεικνύουν ότι οι κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση των οπτικοακουστικών παρόχων έχουν πλέον ουσιαστική σημασία για την μελλοντική ρύθμιση ή απορρίθμιση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας την καινοτομία αλλά και τις υπηρεσίες δημόσιου και οικονομικού συμφέροντος. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα το οποίο ουσιαστικά καλούμαστε να επιλύσουμε. Είναι σαφές ότι η συζήτηση περί κρατικής χρηματοδότησης επικεντρώνεται καταρχήν στους λεγόμενους δημόσιους παρόχους ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών όπως αυτοί ορίζονται από το κάθε κράτος μέλος δεδομένων των ουσιαστικά μικρότερων πόρων που έχουν στη διάθεσή τους αλλά και πρωτίστως του σημαντικού ρόλου κοινής ωφελίας που τους έχουν ανατεθεί. Ο σημαντικός ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών αναφέρονται στη σύμβαση UNESCO, στο πρωτόκολλο Άμστερνταμ αλλά και στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001. Ήδη υπάρχει δηλαδή μία πλατφόρμα όπου ορίζεται σαφώς ο ρόλος των δημόσιων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχει ανοίξει όμως ο φάκελος της συζήτησης των κρατικών ενισχύσεων και θα πρέπει να λάβουμε ορισμένα νέα δεδομένα όπως ορίσατε, αλλά και ορισμένες ενέργειες που δημιουργούνται ή θελημένα ή αθέλητα, λόγω της σύγχυσης η οποία υπάρχει μεταξύ πολλές φορές δημόσιου και ιδιωτικών φορέων θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα ζητήματα. Πρώτο, το θέμα του ορισμού της εντολής δημόσιας υπηρεσίας δεν θα πρέπει να συγχέεται με το θέμα του χρηματοδοτικού μηχανισμού που επιλέγεται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. συνεπώς ενώ η δημόσια τηλεόραση μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες όπως πώληση διαφημιστικού χρόνου προκειμένου να επιτύχει ορισμένα έσοδα. αυτό ορισμένες κυβερνήσεις όπως από τη γαλλική κυβέρνηση έχει καταδικαστεί και ανατρέπεται με βάση την εθνική νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, οι εμπορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που υπόκειται στην υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας διαδραματίζουν και αυτή σημαντικό ρόλο. Η συνύπαρξη ιδιωτικών και δημόσιων παρόχων υπηρεσιών αποτελεί βασικό συστατικό σημείο της ευρωπαϊκής αγοράς. Με ένα ζήτημα, Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω ότι οι προτινόμενες από την επιτροπή εκ προτέρων διαδικασίες εξέτασης των κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να μας προβληματίσουν όχι διότι αναβάλλεται ή επικαλύπτεται η επικουρικότητα αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι συμβατές με τους όρους των κρατικών ενισχύσεων και στο τέλος πρέπει να πούμε ότι το θέμα των εθνικών ενισχύσεων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να εξεταστούν και στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων διότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν να ανταγωνιστούν διεθνώς κολοσσούς και μια αυστηρή νομοθεσία θα βλάψει το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και κοινοτικό κεκτημένο. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Για τους ε, για δύο λεπτά, ο κύριος Ιγνάση Γκουεντάνς Καμπό. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ξεκινώ και εγώ ε, αποστέλλοντας τις καλύτερες ευχές μου για αποκατάσταση της υγείας της κυρίας Κρούς. Ελπίζω να, να, κάψει ε, από την πτώση που είχε η συζήτηση που έχουμε σήμερα το πρωί είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό ο βασικός λόγος ε, της συζήτησης είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να εμπλακεί το Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος της συζήτησης αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε εδώ. Πριν ολοκληρωθεί η ανακοίνωση τη Επιτροπή, θέλουμε να μπορούμε να έχουμε μια πραγματική συζήτηση στην οποία θα εμπλακούμε όλοι εδώ. Γιατί αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο το μοντέλο τηλεόραση που έχουμε, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Ήδη οι τηλεοράσει, όπω γνωρίζουμε όλοι και όπω μάθαμε όταν συζητούσαμε την οδηγία για τι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων, δεν είναι όπω τι γνωρίζαμε στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα επεξεργάζονται. Ε, περιεχόμενο που το περνούν από την πλατφόρμα, γραμμική, γραμμικά ή όχι, πάντως ε, με τον α τρόπο. Και γι' αυτό η δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης δεν είναι αυτή που ήταν αν κάναμε τη συζήτηση δεκαετία του 70 ή του 80. Προφανώ πρέπει να γίνει η συζήτηση από την άλλη μεριά. Είναι σαφέ. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα ω δημόσια υπηρεσία. Όλα δεν συμβαίνει ότι όλα όσα γίνονται με δημόσια κονδύλια έχουν νόημα σε κάποιες τηλεοράσεις ταυτόχρονα και, αυτό προκύπτει, και από αυτό προκύπτει η ανησυχία μας και αυτό το διαπιστώνω και από συναδέλφους η δημόσια τηλεόραση έχει τεράστια σημασία προστασίας της ποικιλομορφία γλωσσικά και πολιτισμικά. Είναι το Ταμείο Συνοχής των κοινωνιών μας που δεν θέλουν να κερδίσουν ούτω ή άλλως και πάση θυσία. Αυτή την ισορροπία πρέπει να την προστατεύσουμε. Να βρούμε νέους τρόπους ε, χρηματοδότησης, να συζητήσουμε τους νέους τρόπους, αλλά να μην θέσουμε σε κίνδυνο κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις κοινωνίες μας, όπως ακριβώς την σημερινή δημόσια τηλεόραση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Για τους πράσινους, η κυρία Τρίπελ. 1,5 λεπτό. αγαπητοί εκπρόσωποι της Κομισιόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η Κομισιόν Μπαρόζο ε, ανήγγειλε ότι ένας από τους βασικούς της στόχους είναι να απελευθερώσει από υπερβολικές διατάξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις στην ε, Ευρώπη, την αγορά. Ας το κάνει λοιπόν, διότι εδώ βλέπουμε α, αυτό που μας έχει υποβληθεί μία, να είναι μια πρόταση υπερβολικής κανονιστικής ρύθμισης αντί για το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι είμαστε υπέρ τη συνύπαρξης αν θέλετε και των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ραδιοτηλεόρασης. Βεβαίως ε, με λύπη διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα και σήμερα που βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή με νέες τεχνολογίες δεν μπορούμε να αγνωρίσουμε βέβαια ε, να μην αναγνωρίσουμε την πρωτοπορία του ιδιωτικού των, των ιδιωτικών φορέων εκεί και το ότι κάποιες δημόσιες, κάποιοι δημόσιοι ε, φορείς είναι δεινόσαυροι ε, στον τομέα αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως ε, θα πρέπει να, στο, να φροντίσουμε αν θέλουμε να προχωρήσουν καλά τα πράγματα να υπάρξει μια ισορροπία και να αναπτυχθούν και οι μεν και οι δε σωστά. Για την ε, Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κ. Μέγερ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση του κοινού για πολλά θέματα και οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές είναι δυνατόν να γίνονται χάρη στις εισφορές του κοινού και τη δημόσια χρηματοδότηση από εισφορές ορισμένων οργανώσεων όπως γίνεται στην Ολλανδία. Εκτός αυτού όμως η, τα κράτη, η δημόσια υπηρεσία εκπομπών πρέπει και να κερδίζουν κάποια χρήματα, πράγμα που κάνουν μέσω της διαφήμισης ή της δημοσίευσης βιβλίων για οπτικοακουστικά θέματα ώστε να δημιουργήσουν ένα καινούριο κοινό πελατών και να μειώσουν το κόστος για τις δημόσιες υπηρεσίες, για το κράτος. Οι ιδιωτικοί σταθμοί όμως δεν κάνουν το ίδιο και γι' αυτό πολλές φορές οι εμπορικοί σταθμοί θεωρούν ως ε, θεωρούν τους κρατικούς ως ανταγωνιστικούς τους και γι' αυτό προσπαθούν να τους κλέψουν κοινό. Τα συμφέροντα λοιπόν του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα εδώ δεν συμπίπτουν. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να συμβιβάσει ασυμβίβαστα πράγματα. Το μέλλον των δημοσίων ε, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών θα αμφισβητηθεί αν δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να έχουν κάποια εισφορά ή κάποιο κέρδος από ιδιωτικές υπηρεσίες. Από την άλλη μεριά η Κομισιόν τελευταία θέλησε να απαγορευθούν οι συνεργασίες ιδιωτών και δημοσίου τομέα ως προς τη χρηματοδότηση τηλεοπτικών σταθμών. Ο κύριος Μαυρομάτης, τρία λεπτά κυρία επίτροπος όπως υπογραμμίζουν οι συνάδελφοι που υπογράφουν την προφορική ερώτηση και όπως αναλυτικότερα αναφέρθηκαν στην δημόσια ακρόαση την περασμένη εβδομάδα στις βρυξέλλες διακεκριμένοι ομιλητές είναι ανάγκη να δούμε όλοι μας την δημόσια τηλεόραση ως ένα μέσο προσφοράς στους πολίτες που σε ένα μεγάλο βαθμό θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις λειτουργίας της. ο δημόσιος διάλογος η ανεξάρτητη αρχή που τους εποπτεύει καθώς και η ποικιλομορφία των προγραμμάτων σύμφωνα με την ιστορία και τον πολιτισμό κάθε κράτους μέλους είναι ανάγκη να προστατευτούν μετά την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του πλήθους των οργανισμών που αναφύονται καθημερινά. στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού βεβαίως είναι ανάγκη η κομισιόν να αναδείξει καινούριου τρόπους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας τηλεόρασης. κατά κύριο λόγο πρέπει να γίνει σαφής ο καθορισμός της δημόσιας αποστολής των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να γίνει καλύτερη εκτίμηση των κρατικών ενισχύσεων αλλά και στον κανόνα της διαφάνειας είναι ανάγκη να μην γίνονται διακοπές ή άσκοπες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις στα κράτη μέλη και τους δημόσιους φορείς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στην αξιολόγηση που η κομισιόν πραγματοποιεί εκ των προτέρων; να καθιερωθούν αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί ελέγχου στο νέο περιβάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. επιπλέον δεδομένου ότι οι δημόσιοι και οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτισμική και γλωσσική πολιομορφία είναι υποχρεωμένοι και όλα αυτά τα μέσα και οι δημόσιοι βέβαια οργανισμοί και η τηλεόραση να παρέχουν προγράμματα ποιότητας και ταυτόχρονα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με άλλους συναφείς φορείς να δίνονται να ανταποκρίνονται θετικά στις προκλήσεις των καιρών μεταδίδοντας γεγονότα παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως οι ολυμπιακοί αγώνες το παγκόσμιο πρωτάθλημα κτλ. κάτι το οποίο σήμερα δυστυχώς τίνει να ανατραπεί από το γεγονός και μόνο ότι οι ιδιωτικοί φορεί, διαθέτοντας περισσότερα χρήματα δεν μπορεί η δημόσια τηλεόραση να ανταποκριθεί στο κόστος. κατά συνέπεια οι πολίτες δεν θα μπορούν να παρακολουθούν και αυτά τα γεγονότα μαζί με τα υπόλοιπα προγράμματα. ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ακόμα ότι οι σημερινέ προσφορέ τη αγορά και τα συμφέροντα των εμπορικών μέσων ενημέρωση, στον καθορισμό του πεδίου αρμοδιότητας και της δραστηριότητας των δημοσίων φορέων ραδιοτηλεόρασης δεν είναι κατά την ίδια εκτίμηση κάτι το οποίο και εμείς απευχόμαστε βεβαίως εκτίμηση η οποία αφορά το γενικότερο συμφέρον με ελάχιστες φυσικά εξαιρέσεις και αυτό η κομισιόν θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ Μανώλη. Δύο λεπτά η κυρία Μπαντία Κοτσέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, και εγώ να συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους ευχόμενη ταχεία ανάδοση της κυρίας Κρούς. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια σε σχέση με την αναθεώρηση της ανακοινώσεως σχετικά με τη, τις ραδιοτηλεοπτικές μετανόσεις. Να σας πω καταρχάς ότι θεωρώ θετική την αναθεώρηση που ξεκίνησε η Επιτροπή εφόσον θα επιτρέψει να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του 2001 στις αλλαγές που επήλθαν και στο τεχνολογικό πλαίσιο και στην κοινοτική ένωμη τάξη. Επίσης, διότι διατηρεί τους βασικούς άξονες της ανακοίνωσης του 2001 που αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή τηλεοπτικών υπηρεσιών, για να εξασφαλίσουν τον πλουραλισμό και την δημοκρατική ποιότητα. Παραπέμπω ιδιαίτερα στις αρχές του ορισμού και περιορισμού από πλευράς κρατών του περιεχομένου και της βάσης της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν αναλάβει οι αντίστοιχες δημόσιες, ε, τα αντίστοιχη ε, ε, ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και να αποφεύγουν την στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα την, για την, ολοκλήρω, την ανάθεση του ελέγχου της αποστολής αυτής μέσω συγκεκριμένης διαμόρφωσης του πλαισίου και την ανεξάρτηση εξάρτηση της αποστολής αυτής με βασικό ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Επίσης θεωρώ θετικό, θετικούς τους εξάντε ελέγχους στην παροχή των νέων υπηρεσιών από πλευράς των δημοσίων φορέων ραδιοτηλεόρασης εφόσον ωστόσο διατηρείται επαρκή ευελιξία που θα επιτρέπει να προσαρμόζεται η κατάσταση κάθε κράτους στην πραγματικότητα του κράτους. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα προσεκτικά το ενδεχόμενα συγκεκριμένες μορφές παροχής που περιλαμβάνονται στο δημόσιο πλαίσιο των οπτικοκουσών μέσων να ε, αποτελούν αντικείμενο αμοιβή ή αντι Παροχή από πλευρά των δικαιούχων. Δεδομένου του οικουμενικού χαρακτήρα που έχουν και καθολικού χαρακτήρα που είχε πάντα η δημόσια τηλεόραση και των κινδύνων αποκλεισμού που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση που αποδεχθούμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότηση. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα σχόλιά μου αυτά. Ευχαριστώ. Gracias, Ευχαριστώ. Η κυρία Βαντερμπουργκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές ότι το θέμα που συζητούμε εδώ είναι η τάση μεταξύ των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν ε, στην κοινωνία μας για σχετικά με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ε, ε και των ε, ε, υπηρεσιών που παρέχονται της ποιότητάς τους. Ε, βεβαίως εδώ μιλούμε για νέες υπηρεσίες, μιλάμε για την, ε, τον κοινοτόμο χαρακτήρα ενδεχομένως κάποιων νέων υπηρεσιών και που μπορεί να έχουν αντίκτυπο και μάλιστα ε, γενικό υπάρχει βεβαίως το γενικό οικονομικό συμφέρον ε, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής του ε, Κοινοβουλίου και ειδικά η, τα, τα μέλη σοσιαλιστές αυτής της Επιτροπής ε, είπαν σχετικά με το γενικό οικονομικό συμφέρον ότι τα προβλήματα εδώ μπορεί να είναι πολλά, ο αντίκτυπος πολύ μεγάλος και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει πρώτα μία ε, απόφαση πλαίσιο ή ορισμός ενός πλαισίου εντός του οποίου θα κινηθούμε μελλοντικά βεβαίως το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει υποβληθεί για διαβούλευση και στο οποίο μπορούν να γίνουν σχόλια μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και θα γίνουν καλό είναι αυτό καλό είναι να γίνουν σχετικές συζητήσεις νομίζω ότι θα βοηθήσουν αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να δούμε ποιος θα αποφασίσει τους κανόνες και ποια είναι η ισορροπία αν θέλετε μεταξύ των συμφερόντων της αγοράς αφενός και των, του δημοσίου αφετέρου εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της αγοράς που αναφέρει και η Επιτροπή και όχι του δημόσιου τομέα. Εκπλήσουμε που τονίζονται ιδιαίτερα κάποια ε, προβλήματα τώρα από κάποιους ενώ ε, πιο πριν συμφωνούσαν μαζί μας για το γενικό πλαίσιο που πρέπει πρώτα να οριστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά την άποψή μας να αποφασίσουμε οτιδήποτε εάν δεν υπάρχει ένα ορισμένο πλαίσιο επαναλαμβάνω την έκκλησή μας λοιπόν για την ε, δημιουργία ενός πλαισίου που ελπίζουμε να επαναφέρει τελικά την ισορροπία υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Ο κύριος Μποσκούτ, δύο, η Μποσκούτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η δημόσια τηλεόραση προστατεύει την πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη. Δεν το είπα εγώ αυτό, η Επιτροπή το λέει και συμφωνώ μαζί της. Είναι σημαντικά, είναι σημαντική λοιπόν η δημόσιοι οπτικοακουστική φορείς για το λόγο αυτό. Πιστεύω ότι δεν μπορεί η λειτουργία των οργανισμών αυτών να καθορίζεται από τις Βρυξέλλες εξ αρχής είναι κάτι που γνωρίζουν καλύτερα και μπορούν καλύτερα να αποφασίζουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε την αύξηση των κανόνων και την επιβάρυνση των κρατών στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την προσφορά. Δεν πρέπει να ε, δεν, μπορούμε, δεν πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ παλαιών και νέου περιεχομένου. Πολλά παλαιά περιεχόμενα, πολλές μορφές παλαιού περιεχομένου εμπλέκονται και στο νέο πλαίσιο. Το ζήτημα δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο από την οπτική γωνία της αγοράς αλλά και από την οπτική γωνία της καθολικής υπηρεσίας, κάτι που ε, δέχεται και η Επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Επιτροπή, στη νέα εκδοχή της ανακοίνωσης οι αρχές που προανέφερα θα υπάρχουν, θα εμφανίζονται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη και την θέσπιση κανόνων για τις υπηρεσίες κοινού συμφέροντος. Επίσης, θα έχει κάποιο ρόλο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Προχωράμε στη διαδικασία Catch the Eye. Όποιος. Πέντε άτομα. Ο κύριος Μαν για ένα λεπτό. Okay, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι και οικονομικός φορέας. Εγώ πήγα στην Ακρόαση την περασμένη εβδομάδα στις ε, Βρυξέλλες στη σχετική και είδαμε ε, ποια είναι η κατάσταση. 22 κράτη-μέλη είναι αντίθετα ε, προς ε, την ε, θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων διότι τα συστήματα είναι διαφορετικά και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε ένα, μία δοκιμασία εξάντε ε, υποχρεωτική ναι, και, να, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ραδιο τηλεοπτικά συμβούλια σε όλες τις χώρες που ε, ποπτεύουν την κατάσταση υπάρχουν οι αρχές ανταγωνισμού εγώ είμαι ε, μέλος ενός ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου για την ΕΣΥ, για το κρατήριο της ΕΣΥ. Κάνουμε τη δουλειά μας, ελέγχουμε την κατάσταση. Έτσι λειτουργεί σωστά ε, μια αποτελεσματική πολιτική. Ε, η κυρία Ρόιτοβα. Ένα λεπτό. οι συνάδελφοι εκείνοι που είπαν ότι η δημόσια στήριξη ε, στους δημόσιους φο... ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ε, χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεως έχουν δίκιο αυτό το λέμε εμείς εδώ και πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ασχοληθεί με τρία θέματα πρώτα πρώτα κεραίες για το θέμα των κεραιών και των κοινών κεραιών για διάφορα κτίσματα. Από την άλλη μεριά στα και αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα νέα κράτη, τα καινουργια κρατη κράτη-μέλη. Δεύτερο θέμα, οι δημόσιες θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός για να εφαρμόζονται καλύτερα οι κανόνες και τα εθνικά ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια θα πρέπει επίσης να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και τέλος... Ζητώ από την Επίτροπο κυρία Βασιλείου να απαντήσει στις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους σας για την ιδιαίτερα καρποφόρα συζήτηση που θα μεταφέρω στην συνάδελφο κυρία Κρούς. Θα προσπαθήσω, ωστόσο, να σχολιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις σας. Το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ τονίζει την ανάγκη να υπάρχει εξισορρόπηση της χρηματοδότησης, της κρατικής χρηματοδότησης και του ανταγωνισμού. Θέλουν τα κράτη-μέλη να είναι πρωτοπόροι στον τομέα αυτό. Αλλιώ θα χρειαστεί να το αναλάβουμε εμεί στι Βρυξέλλε βάσει καταγγελιών. Ο στόχο μα είναι να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, ενώ οι κανόνες της συνθήκης για τον ανταγωνισμό τηρούνται. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να συνεχίσει να ανανεώνει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί. Η Επιτροπή συμφωνεί επί των στόχων αυτών. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα αποφασίσουν πώς θα χρηματοδοτήσουν τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, κάτι που αναφέρει σαφώς το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μπορούν να πειραματιστούν ελεύθερα με νέα σχέδια. Το σχέδιο ανακοίνωσης καθιστά σαφές ότι τα πιλωτικά σχέδια εξαιρούνται των τεστ ανέκαθεν αναγνωρίζαμε τη δυνατότητα να παρέχεται χρηματοδότηση για δημόσια ραδιοτηλεοπτική αποστολή που περιλαμβάνει ένα ευρύ και ισορροπημένο φάσμα προγραμματισμού από προγραμμάτων συγγνώμη, από τους δημόσιους φορείς ραδιοτηλεόρασης. Αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον. Η Επιτροπή θέλει επίσης να εξασφαλίσει μια μίξη δημοσίου και ιδιωτικού. Έχουμε στόχο να παροτρύνουμε τους δημόσιους φορείς να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες για να εξυπηρετήσουν τις πολιτιστικές, δημοκρατικές και οικονομικές ανάγκες τη νέα κοινωνίας. το τεστ του Άμστερνταμ επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρέχουν χρηματοδότηση για νέες υπηρεσίες μέσων στους δημόσιους φορείς. Προστατεύει τη δυνατότητά του να ε, προλαβαίνουν τις εξελίξεις σε ένα ταχεία ε, μεταβαλλόμενο πλαίσιο. Επίσης είναι προς το δημόσιο συμφέρον να υπάρχουν κίνητρα ωστόσο και για τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Η καινοτομία και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντική για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας. Και είναι ξεκάθαρο προφανές ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είναι ελεύθεροι και θα είναι ελεύθεροι να ξεκινήσουν σε εμπορική βάση οποιαδήποτε νέα μορφή παροχής χωρί προγενέστερη αξιολόγηση. Θέλω να σα διαβεβαιώσω κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την διαβούλευση. Θα αναθεωρήσουμε τα το τεστ για να λάβουμε υπόψη τις θεμητές ανησυχίες. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μας να λάβουν υπόψη τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου στην διάρκεια της αναθεώρησης του σχεδίου. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε κυρίε και κύριοι βουλευτές τη συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό προφορικό, προφορική ερώτηση. Προχωράμε στην σύντομη παρουσίαση, στο επόμενο σημείο, σύντομη παρουσίαση ε, 7 εκθέσεων με βάση το άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους εισηγητές να παρουσιάζουν τις εκθέσεις εντάχει. Ξεκινώ